Είχατε έναν άκρο πεπειραμένο πρόεδρο στο πρώτο τμήμα της Συνόδου και τώρα έχετε μία πολύ άπειρη πρόεδρο στο βήμα. Σας παρακαλώ λοιπόν δείξτε λίγη επίοικια στην απειρία μου. Πάντως θα είμαι σκληρή, σας προειδοποιώ. Συνεχίζω λοιπόν και παρακαλώ να με προσέξετε. Για μια τελευταία φορά το λέω, βλέπω ότι εξακολουθούν να συνομιλούν κάποιοι συνάδελφοι. Εγώ συνεχίζω πάντως δυνάμει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης ε, περί εκλογής ε, των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και άρθρο 4 παραγραφο 1 1-4 του κανονισμού σημειώνει το Κοινοβούλιο την εκλογή του κυρίου Χαβιέρ Κάουσο Περμούη με ισχύ από την 15η Ιουλίου 2014. Καλωσορίζω τον συνάδελφο και αναφέρω ότι δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού μέχρι να ε, αληθευτούν τα διαπιστευτήριά του και να δούμε ε, αν υπάρχουν ενστάσεις ε, θα ε, συμμετέχει ως βουλευτής στο Κοινοβούλιο και στα όργανα με πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του με την προϋπόθεση ότι έχει ε, υποβάλει προηγουμένως τη δήλωση ότι δεν ασκεί κάποιο μη συμβατό με την έδρα του βουλευτή καθήκον. Επίσης η ομάδα του ΕΛΚ ζητά τροποποίηση ε, κάποιων μελών σε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Ο κατάλογος των ορισμών θα περιληφθεί στα πρακτικά και αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών θεωρούνται αυτές οι τροποποίησεις και ορισμοί ότι εγκρίνονται. Πέρα των ανακοινώσεων και περνάμε στην έναρξη της σημερινής συζήτησης. Παρακαλώ εκ νέου τους συναδέλφους. Έχουμε